Pan Preda. Takže kolegové, hezké odpoledne. Dnešní denní zasedání pokračuje. Καλησπέρα σας αγαπητοί συνάδελφοι, επαναλαμβάνω τη συνεδρίαση. Πρώτα απ' όλα έχουμε τα χτεσινά πρακτικά. Τα έχετε διαθέσιμα αυτά όπως και το κείμενο. Υπάρχουν αντιρρήσεις. Εάν όχι εγκρίνονται τα πρακτικά. Και μπορούμε να ξεκινήσουμε με το πρώτο σημείο στη μερίσια διάταξη, το οποίο όπως ξέρετε αφορά τις παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δημοκρατίας και του κράτους δικαίου. Πρώτο θέμα είναι η Σρι Λάνκα. Παρακολούθηση της έκθεσης του ΟΗΕ. Πρώτα απ' όλα θα δώσω τον λόγο στον κύριο Μέρφυ τον συντάκτη της έκθεσής μας. Έχετε το λόγο. Στον σκληρό πόλεμο της κυβέρνησης Σριλάνκα κατά των Ταμίλ σκοτώθηκαν τουλάχιστον 40.000 Ταμίλ μέσα σε λίγες εβδομάδες και εκατοντάδες χιλιάδες κρατήθηκαν σε ανοιχτά στρατόπεδα. Ο ΙΕ επιτέλους αναγνωρίζει τα εγκλήματα εις βάρος των Ταμίλ. Δυστυχώ δεν πρέπει να έχουμε ψευδεστήσει πώ θα αλλάξουν οι συνθήκε για του Ταμίλ στη Σρι Μετά τη δημοσίευση Μα είπανε πω ο Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ θα ξεκινήσει διεθνή έρευνα μόνο εάν συμφωνήσει η κυβέρνηση τη Σρι ή εάν το Συμβούλιο Ασφαλείας ζητήσει έρευνα. Δεδομένη τη φύση τη κυβέρνηση αυτή τη χώρα είναι προφανέ πω δεν θα επιτρέψει διεθνή έρευνα. Τονίζει την ανάγκη να κάνουμε εκστρατεία για να ζητήσουμε ανεξάρτητη έρευνα των εγκλημάτων πολέμου και για να ε, έχει να λογοδοτήσει η κυβέρνηση. 18 Μαΐου θα έχουμε ανά τον κόσμο διαδηλώσεις για τη δεύτερη επέτειο αυτού του πολέμου. Χρειάζεται να παλέψουν από κοινού οι Συγχαλέζοι και οι Ταμίλ για να ανατρέψουν αυτό το καθεστώς. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ εγώ κύριε Μέρφη κύριος Φανόρντεν επίσης για ένα λεπτό. Κύριε Πρόεδρε, λυπούμε ακούγοντας ε, απλά και μόνο τον κύριο Μέρφυ ε, που έχουμε αυτή τη συζήτηση σήμερα που προωθείται από εξτραμιστικά στοιχεία της διασποράς των Ταμίλ ε, και ξεχνάμε πράγματα τα οποία έχουν γίνει, τις πολιτικές δραστηριότητες που έχουν αναλάβει και τις εγκληματικές προσόδους. Η έκθεση των Ηνωμένων Εθνών αποτελεί μία αφορμή για τη συζήτηση αλλά λέει ξεκάθαρα ότι το τη χρησιμοποίησε ανθρώπους ως ασπίδα πολλές φορές, έχει στρατολογήσει παιδιά, μέχρι και παιδιά ε, μεταξύ των δυνάμεών της, έχει εκτελέσει άτομα τα οποία ήθελαν να ξεφύγουν από την περιοχή τους και γενικώ έχει οδηγήσει στον εκτοπισμό πολλών ανθρώπων. Βέβαια, σε καμία περίπτωση πρέπει να βομβαρδίζονται άμαχοι, αλλά νομίζω ότι μας βάζει σε ένα πλαίσιο και βλέπουμε ποιος φταίει τελικά. Και αντί η προσπάθεια ε, να αποσκοπεί στη συμφιλίωση των δύο κοινοτήτων είναι κάποια που προσπαθούν να παροτρύνουν και να υποδαβλήσουν ακόμη περισσότερο το μίσος ε, μεταξύ των δύο πλευρών. Η προσέγγιση είναι δόλια, είναι παραγωγική γιατί στρέφεται κατά της ε, κυβέρνησης ε, που έχει όμως παρόλα αυτά ε, συστήσει την έλελασή για να διερευνήσει τα περιπτώσεις εγκλημάτων. Θα έπρεπε να στηρίξω αυτές τις προσπάθειες και το λόγο της Τριλάνκα και όχι να επιτιθέμεθα εναντίον Το Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Κύριοι συνάδελφοι, ας προσπαθήσετε οι υπόλοιποι να τηρείτε το χρόνο που έχετε για να μην μείνουμε μέχρι τις 6 τα απόγευμα εδώ πέρα. Κυρία Ντεκάιζερ, για δυόμιση λεπτά η επόμενη μιλήτρια. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Καταλάβατε από τα πρώτα λόγια τα οποία αρθρώθηκαν εδώ πόσο έντονη γενικά υπήρξε και πόσο θα, θα γίνει έντονη και σήμερα συζήτηση. Δεν συμφωνούμε με όλα αυτά εμείς ως ομάδα. Εμείς είμαστε υπέρ της δικαιοσύνης και της εμφυλίωσης. Δεν θέλουμε σε χώρες όπου υπήρξαν φρικτοί πόλεμοι όπως αυτός που γίνει στη Σριλάνκα αλλά και σε άλλες βέβαια χώρες δεν μπορεί να υπάρξει συμφιλίωση χωρί να αποδοθεί δικαιοσύνη. Η έκθεση των Ηνωμένων Εθνών, κύριε Βαν Όρντεν, σίγουρα περιγράφει κάποια πράγματα. Αναφέρει περιστατικά, αναφέρει γεγονότα και ζητά να καθιερωθεί ένα διεθνή ε, μηχανισμό απόδοση δικαιοσύνη, μέσω βέβαια και τη συμφωνία τη κυβέρνηση. Και αυτό είναι το ελάχιστο. Η ελάχιστη προπόθεση. Πώ θέλετε εσεί να συμφιλειωθεί ο λαό τη Σρι αν δεν γίνει αυτό. Και μιλάμε και για τις δύο πλευρές, δεν μιλάμε μόνο για τους Ταμίλ. Και από τις δύο πλευρές διαπράχθηκαν εγκλήματα και οι δύο πλευρές έχουν ευθύνε και οι δύο πλευρές θα πρέπει να... Ε, και για τις δύο πλευρές θα πρέπει να δοθεί δικαιοσύνη. Δεν έχουμε ε, υψηλά πρότυπα συμφιλίωσης εύκολα όταν έχουμε ένα εθνικό ε, σύστημα δικαιοσύνης γιατί δεν μπορεί να διευκρινίσει ό,τι έχει γίνει. Εγώ νομίζω ότι σήμερα το Κοινοβούλιο όμως το μόνο που μπορεί να κάνει είναι να στηρίξει την έκθεση αυτή για να χυθεί το φως και να, δοθεί, να αποδοθεί δικαιοσύνη. Αυτό είναι το μόνο μήνυμα το οποίο θέλω να μεταφέρω. Ίσως να μην έχω εξαντλήσει και το χρόνο αγόρευσης, αλλά ουσιαστικά έχω ολοκληρώσει. Αυτό ήθελα να πω. Εξαιρετικά, λέει ο Πρόεδρος. Ο επόμενος ομιλητής, Τόμας Μάν. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Το Φεβρουάριο ταξίδεψα με την ε, αντιπροσωπή για την νοτιοανατολική Ασία στη Σρι Λάνκα και είδαμε τις προσπάθειες αντιμετώπισης των συνεπειών ενός 25 ετούς ε, εμφυλίου πολέμου. ΟΗΕ και ΜΚΟ προσπαθούν να απομακρύνουν τις νάρκες για να επαναγκαταστήσουν τους Ταμίλ στη... στόπους όπου έμεναν. Διαπίστωσε ο ΙΕ εγκλήματα πολέμου, εγκλήματα κατά τους, ε, της ανθρωπότητας και από τις δύο πλευρές. Ενθαρρυντικό είναι η σύσταση μιας επιτροπής ε, για την συμφιλίωση και για την ε, αντιμετώπιση των παλαιών πολεμιστών. Οπότε θα πρέπει να υπάρχει η διάθεση ενσωμάτωση των μειονοτήτων και τήρησης των διεθνών προδιαγραφών δικαίου για να αναπτυχθεί αυτή η χώρα χωρίς βία και χωρίς τρομοκρατία. Απευθύνουμε έκκληση στην ύπατη εκπρόσωπο να υποστηρίξει τέτοιες προσπάθειες. Ευχαριστώ πολύ κυρία Μαν. Η κυρία Γιάτεν Μακή. Πρόεδρε, η σύγκρουση στη Σρι Λάγκα μας κάνει να θέτουμε πολλά ερωτήματα τα οποία δεν μπορούμε να απαντήσουμε. Ε, εδώ λοιπόν πρέπει να δούμε ότι χρειάζεται χρόνος, δέσμευση και προσπάθειες, καθώς και ισχυρή βούληση, ώστε να αντιμετωπίσουμε τις πληγές που έχει αφήσει πίσω της η σύγκρουση. Είναι απαραίτητη η συμφιλίωση και η δικαιοσύνη είναι απαραίτητη για να γίνει μια νέα αρχή. Οπότε η κυβέρνηση της Σιλάνκα θα πρέπει αμέσως να αρχίσει τις έρευνες για τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του ανθρωπίνου δικαίου. Και στις δύο πλευρές πρέπει να γίνουν έρευνες. Οι διεθνείς συμβάσεις όπου έχει προσπογράψει η Σρι απαιτούν ακριβώς να γίνουν έρευνες για τις καζόμενες παραβιάσεις και για τους αυτοργούς τους. Μόνο με ανοιχτή και έντιμη έρευνα μπορεί να ξεπεράσει τις πληγές αυτής της δύσκολης και αιματηρή σύγκρουση, ο λαός της Σιλάνκα και να ζήσει σε συνθήκες ειρήνης. Ο Γενικός Γραμματέας ε, του ΟΗΕ με την έκθεσή του, ο κ. Μπανκιμούν, και την πρωτοβουλία αυτή, ε, νομίζω ότι πρέπει να στηριχθεί στην προσπάθειά του με τις συστάσεις μας. Ευχαριστούμε κυρία Χαουτάλα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. 23 Μαΐου 2009 ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, ο Μπανκιμούν και ο Πρόεδρος της Σρι υπέγραψε μια κοινή δήλωση με την οποία συμφώνησε η Σρι σε λογοδοσία για τα εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας κατά τη διάρκεια του πολέμου που τελείωσε το Μάιο του 2009. Μετά από αυτή τη συμφωνία, η οποία δεν τιμήθηκε, δεν τηρήθηκε από την κυβέρνηση της ε, Σρι έστειλε μια ομάδα ειδικών ΟΗΕ για να συμβουλεύσει. Τώρα δημοσιεύτηκε μια έκθεση και βρήκε σοβαρές κατηγορίες πως και οι κυβερνητικές δυνάμεις και οι αντάρτες Ταμίλ δεν σεβάστηκαν το διεθνές δίκαιο. Και τονίστηκε η ανάγκη λογοδοσίας και από τις δύο πλευρές. Ξακολουθεί η κυβέρνηση της Σρι Λάγκας να αποκαλεί την έκθεση αυτή παράνομη και προκατηλημένη. Εγώ θεωρώ πως είναι αντικειμενικός λόγος για περαιτέρω έρευνες σε καιρό που αμφισβητούνται τα έργα των διεθνών οργανισμών, εμείς θα πρέπει να υπερασπιστούμε το διεθνές δίκαιο. Τα εγκλήματα πολέμου δεν πρέπει να μείνουν ποτέ ατιμόρυτα όπου και αν συμβαίνουν. Και τώρα οι ομιλητές των πολιτικών ομάδων. Πρώτα απ' όλα κύριε Κορχόλα για το ΕΛΚ. Ευχαριστώ, Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ο εμφύλιος πόλεμος κράτησε 25 χρόνια με την ήττα των τίγριων, των Ταμίλ και με χιλιάδες θύματα, χιλιάδες νεκρούς. Τελευταίες ε, φάσεις του πολέμου μάλιστα ιδιαίτερα ματηρές με πολλούς ε, αμάχους να χάνουν τη ζωή τους. Και υπάρχουν ε, παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Οι Ταμίλ φαίνεται να έχουν χρησιμοποιήσει ανθρώπινες ασπίδες Βέβαια υπάρχουν κατηγορίες και για τις ε, κυβερνητικές δυνάμεις. Θα πρέπει λοιπόν να μπορέσουμε να, θα, πρέπει να είναι δυνατή μια ανεξάρτητη αντικειμενική έρευνα των περιστατικών. Ίσως κάποιοι να μην τη θέλουν αυτή την έρευνα, ίσως κάποιοι να κολλησιεργούν. Οπότε είναι δύσκολο να διεξαχθεί η έρευνα αυτή. Πρέπει να υπάρχει και από τις δύο πλευρές ε, η απαραίτητη καλή βούληση. Πρέπει να στηρίξουμε λοιπόν τις προσπάθειες των ΗΠΑ, των Ηνωμένων Εθνών, Ευχαριστούμε κυρία Γκόμες για τους σοσιαλιστές και δημοκράτες. Η έκθεση του ΙΕ και του Γενικού Γραμματέα Μπαν Κιμούν δείχνουν ότι αναφέρουν μάλλον τι δεκάδε χιλιάδε θύματα και τα ανθρωπιστικά εγκλήματα που διαπρακτικά στη Σιλάνκα, τα οποία θα πρέπει αυτή τη στιγμή να τα αντιμετωπίσει η κυβέρνηση της Σιλάνκα. Θα πρέπει να γίνει μια ανεξάρτητη έρευνα, να εντοπιστούν οι αυτούργοι, αλλά αυτό δεν είναι θέμα καν πολιτική επιλογή. Είναι μια αρχή που επιβάλλεται από το διεθνέ δίκαιο. Η Επιτροπή Συμφιλίωση που δημιουργήθηκε από την κυβέρνηση δεν καλύπτει σοβαρές βασικέ προποθέσει ανεξαρτησία. Έτσι λοιπόν, το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ καθώ και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να επιμείνουν και να απαιτήσουν μέσω τη έκθεση αυτή τη δημιουργία ενό ανεξάρτητου διεθνού μηχανισμού, ο οποίο να ελέγχει ε, τι ενέργειε τη κυβέρνηση, να ερευνήσει τα εγκλήματα που διαπράχθησαν και από τι δύο πλευρέ και να επιτρέψει ανεξάρτητη απόδοση δικαιοσύνη για το λαό τη Σρι Ευχαριστώ κυρία Μπιλμπάμπορα Ραντίκα εκ των Φιλελευθέρων Δημοκρατών. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να στηρίξω το ψήφισμα για τις παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τα εγκλήματα πολέμου στη Σρι Λάγκα και την αλληλεγγύη μας προς τα θύματα πρέπει να εκφράσουμε και τα βία γεγονότα να καταδικάσουμε, αλλά επειδή δεν υπάρχει ανεξάρτητη δικαιοσύνη πρέπει να στηρίξουμε τη διεξαγωγή μιας αμερόληπτης διαφανούς έρευνας από ανεξάρτητο οργανισμό που θα αποδώσει ευθύνες και θα τιμωρήσει τους ε, αυτούργους. Η ατιμωρησία των εγκλημάτων πολέμου πρέπει να σταματήσει αν δεν θέλουμε να επανειληφθούν τέτοιου είδους ε, επεισόδια. Στη Σρι Λάγκα Μεταξύ άλλων έχουν γίνει βομβαρδισμοί κατά αμάχων. Πριν από 64 χρόνια είχαν ε, ε, βομβαρδίσει οι δυνάμεις του ε, Φράγκο την Κερνίκα. Και αυτό βέβαια έχει αποδοθεί στον πίνακα το γνωστό του Πικάσο που αποτελεί σύμβολο ειρήνης. Αλλά στόχος μας πια είναι να περάσουμε προς την συμφιλίωση. Πρέπει να στηρίξουμε λοιπόν τη Σρι και να απαιτήσουμε την κυβέρνησή τη να εγκαταστρέψει τις διαδικασίες που θα φέρουν στη χώρα ειρήνη και δημοκρατία. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Και τώρα κυρία Ντελή, εκ μέρους των Πρασίνων. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Η έκθεση των Ηνωμένων Εθνών που δημοσιεύτηκε στις 11 Απριλίου του τρέχοντος ε, ρίχνει φως στα εγκλ... τα εγκλήματα πολέμου και τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας στη Σιλάνκα που έφεραν σε αντιπαράθεση τις ε, δυνάμεις τις κυβερνητικές με τους τίγρεις ε, των Ταμούλ. Εδώ λοιπόν, των Ταμίλ μάλλον. Εδώ έχουμε εγκλήματα πολέμου, εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, όπου χιλιάδες πολίτες βρήκαν το θάνατο και δεν μπορούμε βεβαίως να μείνουμε αμέτωχοι και να αφήσουμε τους αυτούργους ε, ατιμόρυτους. Η κυβέρνηση έχει κάνει τα ώστε η έκθεση του ΟΗΕ να μην δημοσιευτεί και αμφισβητεί και τα ίδια τα συμπεράσματά τη, τα πορίσματά τη. Στην Σριλάνκα ο τύπο υπόκειται σε σε λογοκρισία. Υπάρχουν ε, αυθαίρετε συλλήψει και κρατήσει δημοσιογράφων και οι δικαστικές αρχές δεν μπορούν να εκτελέσουν το έργο τους. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει δυνατότητα να πρόσβασης από τον ΟΗΕ και τους υπαλλήλους τους στα, στα δόπεδα των, που βρίσκονται οι πρόσφυγες. Εδώ λοιπόν πρέπει αμέσως να αποσταλεί αποστολή παρατήρησης του Κοινοβουλίου, ώστε να παρακολουθήσει τι συμβαίνει ακριβώ στην ε, Σιλάνκα και να εξασφαλίσει τα ανθρώπινα δικαιώματα και το δικαίωμα αυτοδιαχείριση των λαών. Ευχαριστούμε, η κυρία Βερζιά. Ε, υπάρχει γαλάζια κάρτα τον κύριο Τάνοκ. Θέλετε να... Κυρία Ντελή, θα δεχτείτε το ερώτημα του κυρίου Τάνοκ. Άλλαζε κάρτα. Yes, are you... When we have blue card, you have to say whether you are willing to accept the question. Όταν υπάρχει μπλε κάρτα, γαλάζια κάρτα, πρέπει να πείτε αν δέχεστε ή όχι να απαντήσετε στο ερώτημα. Κύριε Τάνοκ, πρόεδρε, άκουγα στα γαλλικά τι έλεγε ο Μιλήτρια και χρησιμοποίησε τον όρο γενοκτονία, γενοσύντ, που έχει ιδιαίτερο νόημα ω όρο στο διεθνέ δίκαιο. Εδώ όμω ε, η κυβέρνηση πώ ε, μπόρεσε να απελευθερώσει 200.000 ε, που κρατούνταν ω τώρα ως φυλακισμένοι. Είναι δυνατόν να κατηγορείται αυτή η κυβέρνηση για γενοκτονία. Κυρία Ντελή, ακούσατε το ερώτημα. Αν έχετε την καλοσύνη να απαντήσετε, παρακαλώ. Κύριε Βουλευτά, χρησιμοποίησα τη λέξη αυτή που είναι μια μεταφορά ουσιαστικά, αλλά ήθελα κυρίως ε, να περιγράψω το φαινόμενο και είπα ότι δεν είναι το όνομα που χρησιμοποιούμε τελικά. Πρέπει να επαληθεύσουμε. Αλλά αυτά που γίνονται για την μειονότητα τα δεν μπορεί κανείς να τα χαρακτηρίσει ανώδυνα και δίκαια. Thank you. Ευχαριστώ πολύ κύριε Φανόρντεν. Έχετε κι εσείς σηκώσει μπλε κάρτα προς την κυρία Ντελή. Θέλετε, κυρία Ντελή, να δεχτείτε. Ναι, ευχαριστώ πολύ. Η προλαλήσασα. Είπε ότι ζητεί κάποια επιτροπή να συσταθεί, να πάει στη Σιλράνκα να δει όπου τι συμβαίνει. Θέλω να τη υπενθυμίσω ότι η νοτιοανατολική αντιπροσωπεία πήγε πρόσφατα στη Σρι και είναι παρόντες κάποιοι από αυτούς που συμμετείχαν σε αυτή την αντιπροσωπεία. Ο συνάδελφο, ο κύριος Μαν μάλιστα, αναφέρθηκε στην ε, επίσκεψη. Μάλλον δεν ακούει η κυρία Ντελή τι λέγεται στη συζήτηση. Υπάρχει κόσμο που έχει πάει στη Σρι Λάγκα, που ξέρει τη Σρι Λάγκα και που ξέρει τι γίνεται. Αυτέ οι ανοησίε δεν ξέρω από πού τι έχετε βγάλει. Madame Κυρία Ντελή, έχετε δίκιο. Ήδη αποστήλαμε αποστολή στη Σρι Και πραγματικά πρέπει να ήταν θαυμάσια η αποστολή αυτή, αφού και εσεί εργαστήκατε ε, για να πετύχει. Όμω θα πρέπει να ασκήσουμε και πίεση. Πρέπει τέτοιου είδου ε, πρωτοβουλίε να τι επαναλάβουμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Και τώρα, επόμενη ομιλήτρια, κυρία Βερζιά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η Σιλάνκα είναι μια χώρα τραυματισμένη. Ο εμφύλιος πόλεμος θα έχει λήξει πλέον σε λίγο καιρό, εδώ και μια διετία. Και ξέρουμε όλοι πόσα φρικτά πράγματα συνέβησαν. Οι εκθέσεις των μη κυβερνητικών οργανώσεων εδώ είναι απογοητευτικές. Χιλιάδες είναι οι άμαχοι και οι πολίτες που σκοτώθηκαν μέχρι τον ε, Ιανουάριο του 2009. Οι φιλοκυβερνητικές δυνάμεις απέκλεισαν ολόκληρες γεωγραφικές ζώνες και υποτίθεται ότι ενθάρρυναν τους πρόσφυγες να μεταβούν εκεί. Όμως έκτοτε από την φετινή χρονιά προσπαθούν ε, οι κυβερνητικοί της Ιλάκα να άρουν κάθε υποψία εναντίον τους και να εμποδίσουν το ανεξάρτητο έργο της δικαιοσύνης. Οι πολίτες λοιπόν που βρίσκονται στις πρώην περιοχές του εμφυλίου πολέμου δεν, έχουν, δεν μπορούν να λάβουν καμία ανθρωπιστική βοήθεια μέχρι και τρόφιμα ή περίθαλψη. Έτσι λοιπόν ε, τα λάθη αυτά δεν μπορούν παρά να αναγνωριστούν. Έχουν χρησιμοποιηθεί ακόμη και παιδιά στρατιώτε και ανθρώπινε ασπίδε σε αυτόν τον πόλεμο. Θα πρέπει οι κυβερνητικέ δυνάμει που θα αναλάβουν, ε, μάλλον αυτά που προτείνουν τώρα οι κυβερνητικέ δυνάμει δεν δικαιολογούν τη σημερινή απραξία. Η κυβέρνηση τη Σιλάνκα αυτή τη στιγμή έχει επαναλάβει του ελιγμού τη για να εμποδίσει τη δημοσίευση, ιδίω τη τελευταία έκθεση και να απορριφθούν τα πορίσματά τη. Δεν μπορούμε λοιπόν παρά να εκφράσουμε την ικανοποίησή μα για την έκθεση τη 11η Απριλίου. Η σύσταση που σήμερα μα υποβάλλεται ε, οδεύει προ τη σωστή κατεύθυνση. Εγώ θα θέλω όμω να πηγαίνει και λίγο μακρύτερα. Διότι πραγματικά ήρθε η στιγμή ώστε η διεθνή δικαιοσύνη να περάσει και από τη Σιλάνκα όπω έχει κάνει κι αλλού. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Πάσκα για την Ευρώπη της Ελευθερίας και της Δημοκρατίας. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, η σύγκρουση που διήκησε δεκαετίες μεταξύ ανταρτών Ταμίλ και της κυβέρνησης της ε, Σρι Λάγκα ε, επιτέλους τελείωσε το 2009. Μετά το τέλος της σύγκρουσης ο πρόεδρος της ε, Σρι Λάγκα υποσχέθηκε να ερευνήσει όλες τις καταγγελίες παραβίασης του στρατιωτικού δικαίου και του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου. Η έκθεση του ΟΗΕ που δημοσιεύθηκε τον Απρίλιο λέει πως και οι δύο πλευρές ε, διεξήγαγαν στρατιωτικές επιχειρήσεις χωρίς να προστατεύσουν ζωές και δικαιώματα των πολιτών. Παρ' όλα αυτά, οι κρατικές αρχές δεν μπόρεσαν να ερευνήσουν ε, τα γεγονότα και να υπάρξει κάποια λογοδοσία. Πρέπει να υποστηρίξουμε την προσπάθεια του ΟΗΕ για να υπάρξει κράτος δικαίου Σρι Λάνκα και λογοδοσία για δολοφονίες και ακροτηριασμούς χιλιάδων πολιτών στην Σρι Λάνκα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Κατσμάρεκ έχει τον λόγο. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, τα δραματικά γεγονότα της ε, Σρι Λάνκα που περιγράφονται στην έκθεση του ΟΗΕ δείχνουν σαφώς ε, τι προβλήματα μπορούν να δημιουργηθούν από μια στρατιωτική σύγκρουση. Αυτό το οποίο συνέβη είναι απόδειξη του ότι αν προσπαθούμε να δημιουργήσουμε τα προβλήματα με το στρατό θα τα κάνουμε χειρότερα. Για πολλά χρόνια ε, μιλάει ο κόσμος για το λεγόμενο δίκαιο πόλεμο αλλά δυστυχώς στο σημερινό κόσμο οποιοδήποτε πόλεμος, ακόμα και αν θεωρητικά είναι δίκαιος, θα έχει θύματα αθώα. Αν ξέρετε του πώς τα ορίζουμε. Στην περίπτωση της Σρι Λάγκα φαίνεται ότι ο πόλεμος δεν ήταν δίκαιος για κανέναν. Δεν έχει πάντα δίκαιο νικητής, αν και αυτό προσπαθεί να αποδείξει. Εάν είναι να υπάρξει συμφιλίωση, όπως λέει η κυβέρνηση, αυτή πρέπει να βασίζεται στην αλήθεια για το τι συνέβη κατά τη διάρκεια του πόλεμου. Δεν θα υπάρξει αληθινή συμφιλίωση αν δεν αποκαλυφθούν τα εγκλήματα πολέμου ανεξαρτήτως του ποιο τα διέπραξε. Δεν θα υπάρξει συμφιλίωση εκτός εάν τα μέρη αντιληφθούν πως δεν υπάρχουν ταμπού. Όσον αφορά τι αμαρτίε του, θα δώσω τώρα τον λόγο στον Κλοντ Πρόεδρε, πολλοί είναι όσοι στην Ολομέλεια αυτή έχουν αναμειχθεί στις πολιτικές ε, υποθέσεις της Σιλάνκα και στη διασπορά τη Σιλάνκα και τη κοινότητα των Ταμίλ. Αυτό που συζητούμε σήμερα είναι μια έκθεση του Γενικού Γραμματέα και του πάνελ επιρογνωμόνων ε, για την αξιοπιστία τη Σιλάνκα. Δεν άκουσα κανένα στην ε, αίθουσα τη Ολομέλεια ακόμη να εκφράζει αμφιβολίε για την ακαιρεότητα και την εντυμότητα με την οποία έχει συνταχθεί η έκθεση αυτή. Εγώ διαβάζοντα την έκθεση Μπορώ να πω ότι υπάρχουν επικριτικά σχόλια και για τις δύο πλευρές. Θα πρέπει λοιπόν να αφήσουμε την έκθεση αυτή όπως έχει, να δούμε κατά πόσον οι έρευνες χρειάζονται από τον, για τα όσα συνέβησαν από τον Ιανουάριο μέχρι τον Απρίλιο. Και νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό το Διεθνές Φόρουμ των Ταμίλ να ληφθεί υπόψη στην έκφρασή του για το ότι θα πρέπει και οι δύο πλευρές να ερευνηθεί τι σφάλματα διέπραξαν, ιδίως ε, για τη στάση του LTT. Εδώ χρειαζόμαστε δικαιοσύνη, συμφιλίωση και μια επώδυνη έρευνα που μπορεί όλους να τους ε, ενοχλεί, παρόλα αυτά θα πρέπει να την φέρουμε εις πέρας. Ευχαριστούμε κύριε Μωράης και κυρία Αντρικένε. Κύριε Πρόεδρε, είναι αποτροπιαστικό ότι στη διάρκεια της μακράς στρατιωτικής συγκρούσης στη Σριλάκα, η οποία έληξε το 2009, Σχεδόν 100.000 ε, άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, μεταξύ των οποίων δεκάδες χιλιάδες άμαχοι που πέθαναν έχασαν τη ζωή τους στη τελευταία φάση των συγκρούσεων. Η διεθνής κοινότητα θα πρέπει να απαιτήσει να γίνει μια έρευνα ανεξάρτητη η οποία θα διερευνήσει τους αποτροπισμούς που έγιναν και τις φρικαλότητες που έγιναν και από τις δυο πλευρές. Υπάρχουν χώρες όπως η Ρωσία που δεν συμφωνούν να γίνει συζήτηση σε επίπεδο εθνών. Ο Γενικό Γραμματέα του ΕΕ θα πρέπει να είναι πιο αποφασιστικό και να ζητήσει τη διεύνηση των εγκλημάτων πολέμου. Η έκθεση των υπερογνωμών του ΟΗΕ αναφέρει σαφεί παραβιάσει ε, του νόμου περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων ε, από την κυβέρνηση τη Σριλάνκα αλλά και από του αντάρτε Ταμίλ. Κάποιοι από αυτές, κάποιες από αυτές τις δράσεις θα μπορούσαν να θεωρηθούν εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, ε, εγκλήματα πολέμου. Θα πρέπει λοιπόν να συγκροτηθεί άμεσα ο μηχανισμός δικαιοσύνης που προτείνει και η έκθεση του ΟΗΕ. Ευχαριστώ. Thank you. Σας ευχαριστούμε και τώρα θα περάσουμε στη διαδικασία προσέλκυσης προσοχής του Προέδρου. Διαδικασία Catch the Eye. Δύο ομιλητές μπορούν μόνο να πάρουν το λόγο. Έχω δέκα παρόλα αυτά εγγεγραμμένος. Τέσσερις ε, θα μπορέσουν να μιλήσουν τελικά. Κυρία Εσάια είναι η πρώτη. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, στην έκθεση των Ηνωμένων Εθνών είναι σαφές, όπως λέγεται τουλάχιστον, ότι η σύγκρουση αυτή που διήρκεσε 25 χρόνια είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους σε μεγάλος αριθμός αμάχων. Και στα χέρια των ε, κυβερνητικών δυνάμεων αλλά και στα χέρια των ανταρτών ταμίλ με δολοφονίες, με τη χρησιμοποίηση στους ανθρώπινες ασπίδες. Έχει πραγματικά παραβιαστεί το διεθνές δίκαιο, τα ανθρώπινα δικαιώματα. Τώρα έχουν ξεκινήσει κάποιες ε, διαπραγματεύσεις και ίσως θα ήταν καλό υπό την αιγύρια των ΗΠΑ να ξεκινήσει ταυτόχρονα και μια ανεξάρτητη έρευνα. Η πρότασή μας είναι ισορροπημένη και μένουμε ακριβώς αυτό στην ανάγκη να συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις και να υπάρξει συμφιλίωση. Κούτας, επόμενος ομιλητής. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Τα συμπεράσματα της έκθεσης του ΟΗΕ που δημοσιεύθηκε στις 25 Απριλίου είναι σοβαρές κατηγορίες για πολλαπλές παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και διεθνούς δικαίου από την κυβέρνηση της Σριλάνκα και τις επαναστατικές δυνάμεις που ιτήθηκαν στην εμφυλία σύγκρουση που διήρξε πάνω από 25 χρόνια και σκοτώθηκαν δεκάδες χιλιάδες ε, πολίτες από βομβαρδισμούς νοσοκομείων ακόμα και κέντρων του ΟΗΕ. Από την άλλη, οι επαναστάτες χρησιμοποίησαν ανθρώπους ως ανθρώπινες ασπίδες και όσοι προσπάθησαν να φύγουν ε, πυροβολήθηκαν επί τόπου. Οπότε σημαντικό είναι να υπάρξει ένας ανεξάρτητος διεθνής μηχανισμός για να ερευνήσει τα εγκλήματα πολέμου σε αυτή την χώρα. Χρειάζεται μια μερόληπτη έρευνα διαφανής για να ξεχαρίσει ποιος είναι υπεύθυνος για αυτά τα εγκλήματα. Ευχαριστώ, Γκράιμ Βάτσον. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Η μελετημένη αυτή η έκθεση μας δείχνει πέρα από όλα τα συμπεράσματα πως η πρώτη απώλεια κάθε πολέμου είναι η αλήθεια. Αυτό το οποίο δεν κάνει είναι να λέει ποια πολιτική θα πρέπει να γιατρέψει τις πληγές αυτής της χώρας. Πάρα πολλές χώρες για πολύ καιρό κάνουν τα στραβά μάτια, ε, έκαναν τα στραβά μάτια στο τι συνέβαινε. Τώρα πρέπει μέσω μιας συντονισμένης προσπάθειας της διεθνούς κοινότητας να ε, προσπαθήσουμε να βρούμε δικαιοσύνη για όλους όσους έχουν τόσο φοβερά επηρεαστεί. Είστε Ρωμέβα Ιρουέντα. Ρωμέβα Ιρουέντα είναι ο επόμενος ομιλητής. Ευχαριστώ. Ο κύριος Γότσον το είπε και αυτός, ότι το πρώτο θύμα ε, στον πόλεμο είναι ακριβώς αυτό που είπατε κύριε Γότσον, η αλήθεια. Πρέπει να παραδεχθούμε επίσης ότι το ίδιο το θύμα ή ε, τα θύματα μάλλον τέτοιων συγκρούσεων είναι ο άμαχος πληθυσμό. Και γνωρίζουμε ότι υπάρχουν ευθύνες και για τις δύο πλευρές, κυρίως θα έλεγα ε, και συγκεκριμένα η κυβέρνηση, αλλά και η, η Ταμίλ, LTTE. Πρέπει να γίνει λοιπόν μια έρευνα και θα είναι τα αποτελέσματά της καλά αν η Επιτροπή που θα διερευνήσει τα ε, γεγονότα δεν θα προέρχεται από την κυβέρνηση. Ζητάμε να είναι ανεξάρτητη η Επιτροπή για να διερευνήσει τους ισχυρισμούς που έχει αναφέρει στην έκθεσή της η, ομάδα αυτή του ΟΗΕ. Αλλιώς δεν θα έχουμε λύση. Η ειρήνη θα έρθει αν υπάρχει δικαιοσύνη. Και η δικαιοσύνη είναι δυνατή μόνο εάν είναι βασισμένη στην αλήθεια. Και η αλήθεια θα προκύψει μόνο αν η έρευνα είναι εξάρτητη. Ευχαριστώ. Τελευταίος ο μιλητής, Τάνοκ. Η Στριλάνκα μετά από 25 χρόνια ε, εξεργέσεων και τρομοκρατίας επιτέλους ε, ζει την ειρήνη και υπάρχουν ε, πολλές κατηγορίες των ταμίλ, οι οποίες δεν βασίζονται όμως σε αποδεικνυόμενα στοιχεία. Το θέμα είναι ότι πρέπει να διδαχθούμε από τα να, να αντλήσουμε διδάγματα και ε, να αφήσουμε την Επιτροπή Συμφιλίωση να κάνει τη δουλειά της. Σίγουρα πρέπει να τιμωρηθούν οι ένοχοι για του θανάτους αμάχων. Δεν μπορούμε να θεωρήσουμε ότι αυτά είναι η σκόπιμη κυβερνητική πολιτική. Θέλω να σας πω ότι και το LTT δεν δέχθηκε ε, την ε, προσφορά να παραδοθεί και προτίμησε ένα λουτρό αίματος. Αυτό είναι αποτροπιαστικό. Τώρα υπάρχει μια αμφιθυμία απέναντι στη Σρι Λάγκα, ασκούνται πολλές επιρροές ε, και δεν είναι εύκολο να ε, χαραχθούν εξέλιξη. Η Κίνα τώρα προσπαθεί να γεφυρώσει κάποιο χάσμα και να γίνει ο μεγαλύτερος φίλος της Σρι Λάγκα στο πλαίσιο του ΟΗΕ, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε το δικό της ιστορικό σε ό,τι ανθρώπινα δικαιώματα. Ευχαριστώ. Θα δώσω τώρα το λόγο στον Επίτροπο, τον κύριο Άντορ, για να μας δώσει την άποψη της Κομισιόν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Στις 25 Απριλίου 2011, τα Ηνωμένα Έθνη δημοσίευσαν τη συμβουλευτική έκθεση του πάνελ επιγνωμόνων που ε, προσυπέγραψε και ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ σε σχέση με την λογοδοσία και την ένοπλη σύγκρουση βεβαίω στη Σρι Ε, η ομάδα εμπειρογνωμόνων θεώρησε ότι είναι βάσιμε κάποιε από τι κατηγορίε ε, σε σχέση με τι συνεχεί παραβιάσει των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, του διεθνού δικαίου για τα ανθρώπινα δικαιώματα από τον στρατό τη Σρι και τον στρατό των ε, τη απελευθέρωση των Ταμίλ. Ε, πολλά εγκλήματα μάλιστα συγκεκριμένα κατά της ανθρωπότητας. Οι εμπειρογνώμονε και ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ ε, σύμφωνα με τα λόγια του ΟΗΕ θα πρέπει να καταρτήσουν ένα πλαίσιο μαζί με την κυβέρνηση ε, της Σιλάνκα για την λογοδοσία. Θα πρέπει να ξεκινήσουν έρευνες από την κυβέρνηση της Σιλάνκα σύμφωνα με την έκθεση και να δημιουργηθεί ένας ανεξάρτητος διεθνής ε, ε, μηχανισμός για το σκοπό αυτό από το Γενικό Γραμματέα. Επίσης, λέγεται ότι τα πορίσματα της έκθεσης ε, μελετώνται από το Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, ενώ ο ύπατος πρόσωπος για τα ανθρώπινα δικαιώματα καλεί την ε, κυβέρνηση τη Σρι Λάγκα να λάβει υπόψη τα πορίσματα σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα και να εξασφαλίσει τη δικαιοσύνη. Η κυβέρνηση όμω τη Σρι Λάγκα απέρριψε την έκθεση αυτή με πολύ δρεμεί όρου. Η ύπατη εκπρόσωπο Κάθριν Άστον δημοσίευσε στην αρχή τη εβδομάδα μια δήλωση εκ μέρου τη Ευρωπαϊκή Ένωση, επαναλαμβάνοντα τι απόψει τη ε, Ευρώπη. Ότι δηλαδή μια ανεξάρτητη διαδικασία για να ε, ερευνηθούν αυτέ οι πολύ σοβαρέ κατηγορίε είναι απαραίτητε για να ενισχυθεί διαδικασία συμφιλίωση και να εξασφαλιστεί η διαρκή ειρήνη και η ασφάλεια στη Σρι Λάγκα. Η ύπατη εκπρόσωπο τονίζει ότι το θέμα τη λογοδοσία θα πρέπει να θεωρηθεί ανασπόσπαστο μέρο τη διαδικασία εθνική συμφιλίωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν ελπίζει ότι η κυβέρνηση της Σιλάνκα θα αναγνωρίσει ότι ο στόχος της έκθεσης αυτής είναι επικοδομητικός. Ενθαρρύνει την ε, συμμετοχή του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ ε, στην ε, υλοποίηση των συμπερασμάτων. Σας ευχαριστούμε, Επίτροπε. Συνάδελφοι, κλείνει η συζήτηση για τη Σρι Λάγκα. Θα ψηφίσουμε μετά την συζήτηση και των υπόλοιπων ε, ψηφισμάτων. Επόμενο θέμα στην ημερήσια διάταξη το Αζερβαϊτζάν. Και δίνω το λόγο στην κυρία Βεζιά. Κύριε Πρόεδρε, δεν συνηθίζω να μιλώ πρώτη και